Okay, we will do what we did last time. Λοιπόν, θα κάνουμε όπως την προηγούμενη φορά που ήταν πολύ αποτελεσματική η ψηφοφορία. Δηλαδή θα μετράω από το 10 μέχρι το 0 και στο 0 θα αρχίζουν οι ψηφοφορίες. Λοιπόν, ελληνικά όμως. Αλλά μετράτε κι εσείς με το μυαλό σας. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επ της έκθεσης του κυρίου Μπέγκε σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εξετάζουμε την πρόταση ψηφίσματος. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 με ονομαστική κλίση. Άρη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 467 ψήφους. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απογύπτεται, as Mr. Schultz said. Απογύπτεται. Τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση. Άρκετη η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα ο κύριος Μάρτιν ζητά το λόγο. Κύριε Μάρτιν, παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίσαμε την τροπολογία υπαριθμών 8. Εμείς όμως Βλέπαμε στην οθόνη ακόμα 7. Θα ήθελα να είναι η σωστή χρονική αλληλουχία και στην οθόνη όπως και αυτές που αναγγέλλεται οι ψηφοφορίες. Παρακαλώ. Λύση. Επομένως ε, αυτό που θα καταγραφεί προφανώς είναι το, το 8. Το 7 το ψηφίσαμε ω χειρός. Ο κύριος Μακμίδαν Μόν θέλει τον... Ε, ορίστε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν λειτουργήσε η ηλεκτρονική μου κάρτα. Αμέσω να σας εξυπηρετήσει. Προχωράμε τώρα στην τελική ε, ψήφο του ψηφίσματος η οποία απαιτεί qualified majority με ονομαστική κλίση άρκετη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. εγκρίνεται με 531 ψήφους. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπέγκε. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης της κυρίας Χάουγκ σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθμός 10-2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009. Μοναδική ε, ψήφος με ονομαστική κλείσει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 559 ψήφους. Συγχαρητήρια στην κυρία Χάουγκ. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης του κυρίου Λένε σχετικά με τον έλεγχο της εντολής. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Λένε. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με συγχωρείτε. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία των πέντε προτάσεων ψηφίσματο σχετικά με τι προοπτικέ για την αναπτυξιακή ατζέντα τη Δόχα, σε συνέχεια τη 7η Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τροπολογία 11. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 563 ψήφους. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Θέλω να το ελέγξω. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 1. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται με 358 ψήφους. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Ε, καταπίπτει, με συγχωρείτε. Τροπολογία 2. Amendment 2. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ο κύριος Ντεζίρ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να δηλώσω ότι αν κατάλαβα καλά την τροπολογία του κυρίου Παπαστάμκου ζητάει να καταργηθούν οι επιχορηγήσεις προς τις εξαγωγές λόγω μιας ε, όμως ενός λάθους που έγινε στο κατάλογο ψηφοφορίας εμείς υπερψηφίζουμε τελικά. Τροπολογία 5 με ονοματική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 326 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 12 σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 13 του αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας εγκρίνεται με 377 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 15. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Το ξανακάνω. Τροπολογία 15. Amendment 15. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 σε δύο μέρη και τα δύο με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 366 ψήφους. Κατά. Δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται με ε, εγκρίνεται με με 493 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 8 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 351 ψήφους κατά. Πάμε λοιπόν στο αρχικό κείμενο της παραγράφου 14 σε δύο μέρη με ονομαστική κλίση και τα δύο. Πρώτο μέρος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται με 574 ψήφους υπέρ. Δεύτερο μέρος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται με 360 ψήφους υπέρ. Η τροπολογία 14 απεσύρθη. Τροπολογία 10 με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται με 364 ψήφους κατά. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 18 ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές ε, να το ελέγξουμε παρακαλώ αρχικό κείμενο παραγράφου 18 Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 358 ψήφους. Και τώρα πάμε στην τελική ψήφο επί του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της οφορίας. Εγκρίνεται με 370 ψήφους υπέρ, 125 κατά και 125 αποχές. Τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. Αλλά προσοχή. At 12 o'clock we have the Zakharov Prize. Έχουμε τώρα το βραβείο Σαχάροφ προχωρήσαμε με μεγάλη ταχύτητα. Τώρα θα πάω πάρα πολύ αργά για να μην φύγει κανείς από την αίθουσα. Και καμία. Προβλέπει την ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων. Μετά την παράγραφο 5 έχουμε δύο τροπολογίες παρομοιότυπες, τροπολογία 1 και τροπολογία 2. Θα τις ψηφίσουμε σε δύο ξεχωριστά μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Θα κάνω ηλεκτρονικό έλεγχο. I will check. Άρχεται η ψηφοφορία. I have to make a phone call if you don't mind. Θα έχω να κάνω ένα τηλέφωνο, με συγχωρείτε μια στιγμούλα. Πρίας. Εγκρίνεται με 502 ψήφους υπέρ. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. This I have to check. Πρέπει να το ελέγξω. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 272 ψήφους κατά. Πάμε τώρα στο αρχικό κείμενο της παραγράφου 11. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνεται και τέλος no, it's και τέλος η ψήφος η τελική ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνεται παρακαλώ όλους συναδέλφους να παραμείνουν στην αίθουσα για το πολύ σημαντικό βραβείο Ζαχάροφ το οποίο θα απονεμηθεί σε περίπου 7 με 8 λεπτά. Και τώρα προχωράμε σε αιτιολογήσεις ψήφου. Για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ο κύριος Μπρεζίνα. Είναι παρόν ο κύριος Μπρεζίνα. Καταψήφισα την έκθεση